δημοκρατικό έθνος και δεν θέλουμε να παίρνουμε μαθήματα από κανένα στη δημοκρα... για τη δημοκρατία και ιδιαίτερω από χώρε που έχουν πολλά να κάνουν οι ίδιες στη χώρα, στο εσωτερικό τους. Ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλδημοκράτες και σοσιαλιστές, ε, Λόπες Αγκουλάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.